Dear colleagues, we can... Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε την κοινή μας συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην κοινή αυτή συνεδρίαση ΕΝΒΙ και ΑΦΕΤ. Θα εξετάσουμε σήμερα τις 369 τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στην κοινή μα έκθεση όσον αφορά την ολοκληρωμένη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αρκτική. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε μια κοινή δήλωση με την ύπατη εκπρόσωπο όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, τι κλιματικέ αλλαγέ και την ειρηνική συνεργασία στην περιοχή τη Αρκτική. Οι προτεραιότητε αυτέ συνάδουν με τι περισσότερε προτεραιότητε για την περιοχή τη Αρκτική που έχει προβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που προωθούν τα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται στην περιοχή τη Αρκτική. Χαίρομαι πάρα πολύ που το σχέδιο έκθεσης, οι τροπολογίες, αλλά πιστεύω και οι συμβαστικές τροπολογίες, επικεντρώνονται ακριβώς τα σημαντικότητα αυτά ζητήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την περιοχή της Ραπτικής. Να δώσω τώρα το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Μπροκ, ο οποίος θα μας πει και αυτός κάποια εισαγωγικά λόγια. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και συμφωνώ απόλυτα με την εισαγωγή που κάνατε. Πιστεύω ότι πρόκειται Όντω ε, για ένα θέμα το οποίο δεν έχει μόνο περιβαλλοντική σημασία, αλλά και όλο ένα και πιο μεγάλη στρατηγική σημασία. Και σε ό,τι αφορά τις νέες δυνατότητες που ανοίγουν από οικονομικοπολιτικής πλευράς, αλλά και για θέματα τα οποία άπτονται των πρωτονυλών. Και άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή η συνδιοργάνωση τις σα. και θα πρέπει τα στρατηγικά μας συμφέροντα να τα λάβουμε υπόψη και από τις δύο σκοπιές. η επιθυμία η οποία εκφράσατε, η περιοχή αυτή να διακατέχεται από περιορισμένε τριβέ και εντάσεις, δεν θα επαληθευτεί. Γνωρίζουμε παράλληλα ότι Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και για τα δικά μας συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα να δώσουμε το λόγο στους δύο εισήγητες. Ο κ. Πάιτ πρώτος. Ε, ευχαριστώ. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, Δυστυχώ ε, η κυρία Πιετικάνη, η συνεισηγητριά μου δεν είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω όμω και αυτήν και του συναδέλφου τη για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε κατά την εκπόνηση τη έκθεση αυτή. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω όλου του κοιόδου συζητητέ για την πολύτιμη και επικοδομητική συμβολή του και στάση του όταν συζητήσαμε τι τροπολογίε. Έχουμε, όπω είπατε, 369 στον αριθμό τροπολογίε, βάσει των οποίων ε, καταλήξαμε σε 21 συμβαστικές προτάσεις, 21 συμβαστικές προτάσεις. Πρόκειται για μια κοινή ε, έκθεση μεταξύ ΑΦΑΤ και ΕΝΒΗ, η οποία ε, εξετάζει τις κλιματολογικές συνθήκες και την αυξανόμενη πρόσβαση στην Αρκτική, καθώς και ενδεχόμενες προκλήσεις στην περιοχή. Αυτό που προσπαθούμε ουσιαστικά να πετύχουμε με την έκθεση αυτή είναι να απαντήσουμε στο σημείο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αρακτική και τα θέματα τα οποία επεξεργάζονται. Αλλά επίση ε, φέρουμε και ευθύνη να πραγματευτούμε και να αντιμετωπίσουμε θέματα τα οποία δεν πραγματεύεται η κοινή ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω είναι η ΚΕΠΑ. Η Αρακτική εδώ και καιρό είναι μια περιοχή επικοδομητική ε, διεθνού εργασίας και έχει χαρακτηριστεί από χαμηλέ συντάσει. Και αυτό θέλουμε να συνεχιστεί. Θέλουμε η Αρκτική να παραμείνει μια περιοχή χαμηλών εντάσεων. Θα πρέπει να μην υπάρξει στρατηγικοποίηση τη περιοχή, ε, να γίνεται σεβαστό το διεθνέ δίκαιο επίση στην Αρκτική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και σημειώνονται ότι η Ρωσία δραστηριοποιείται πιο πολύ στην περιοχή της Αρκτικής και ότι θα πρέπει να συνεχίσει η συνεργασία με την Ρωσία για να παραμείνει ακριβώς ε, σε χαμηλό επίπεδο οποιαδήποτε ένταση στην Αρκτική και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στην Αρκτική και αλλά και άλλα έχουν δικέ του στρατηγικέ. Ε, μεταξύ άλλων ε, και μία διάσταση ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει πιο συνεχτική ιστορική και εξωτερική πολιτική για την Αρκτική και μία στρατηγική και ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράση για την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να ληφθούν υπόψη όλες οι πτυχές, μεταξύ άλλων και η πτυχή της ασφάλειας, αλλά και οι οικονομικές ε, και ενεργειακές εξελίξεις. Και φυσικά ένα από τα σημαντικά στοιχεία της έκθεσης είναι, μεταξύ άλλων, η ηθική και πολιτική αλληλεγγύη με τους αυτόχθονες της περιοχής. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω όλους σας για την καλή συνεργασία. Ελπίζω δε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποδεχθεί την έκθεση αυτή. Σε δύο μήνες ελπίζω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος και ο κύριος Φαρία, ο οποίος ε, θα μιλήσει εξ να της ναι, ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί μου ζητήθηκε από τη συνάδελφο Σύπα Πιετικάινεν που είναι η άλλη εισηγήτρια του ΕΛΚ για αυτό το θέμα και που δεν μπορούσε να είναι σήμερα παρούσα, να σας διαβάσω τις παρατηρήσεις σας. Τις. Ιδού λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτον, Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδελφούς που συνέβαλαν στην σύνταξη του σχέδιου έκθεσης για την ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης ε, Έχαμε καλή συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές ε, από και τις δύο επιτροπές, ε, πράγμα για το οποίο είμαι ευγνώμων. Ε, το περιβάλλον θα πρέπει να συντηρηθεί στις βασικές προτεραιότητες της περιβαλλοντικής ατζέντας της Ένωσης. Οι αλλαγές συμβαίνουν εκεί σε ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αλλού στον κόσμο. Ε, με χαρά παρατήρησα ότι υπήρξαν πολλές παρατηρήσεις από τους συναδέλφους που τόνισαν ε, τις ρήτρες προστασίας του Αρκτικού. Η προστασία του περιβάλλοντος της Αρκτικής, ε, οι διεθνείς συμφωνίες και η σωστή εφαρμογή τους είναι σημαντικός τρόπος να προχωρήσουμε και ο μόνος τρόπος. Η Ένωση πρέπει να παίξει δραστήριο ρόλο στα διεθνή φόρα όπως το ΑΕΜΟ όταν συζητείται η απαγόρευση της χρήση βαρέων καυσίμων όταν πρόκειται για θαλάσσιες μεταφορές στην Αρκτική. Θα πρέπει επίσης να γίνεται ε, η αξιολόγηση επιπτώσεων στον, αρκτικ, αρκτικό κύκλο όταν πρόκειται για σχετικά προγράμματα, πράγμα που θα λαμβάνει υπόψη και τις επιπτώσεις στους ε, ηθαγενείς λαούς. Είναι πολύ σημαντικό να εισακούγονται οι απόψεις τους και να λαμβάνονται υπόψη σε λήψη αποφάσεων που αφορούν τον αρκτικό ε, κύκλο. Πολλοί συνάδελφοι ζητούν ισχυρότερες ε, δικλείδες ασφαλείας για τα δικαιώματα των ε, αυτοχθόνων και αυτές οι προτάσεις έχουν μπει στις συμβιβαστικές τροπολογίες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Γκάλερ εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές και τους σκιώδεις ε, για την επικοδομητική τους εργασία μέχρι στιγμής για τις συμβιβαστικές σας για αυτή την έκθεση. Από την άποψη της εξωτερικής πολιτικής ε, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι δεν πρέπει να επιβαρυνθεί εξαιρετικά αυτό το έγγραφο που θα είναι μια κοινή θέση των δύο επιτροπών μας με τις περιβαλλοντικές πτυχές. Ο τίτλος είναι «Ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον ε, Αρκτική». Και ε, το συζητήσαμε αυτό και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και πολύ αμφιβάλλω ότι όταν έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε οποιαδήποτε περιοχή ή χώρα ως Ένωση δεν θα πρέπει να κλείνουμε προς μια συγκεκριμένη επιτροπή. Η Επιτροπή της Αλίας θα μπορούσε να έχει πει τις δικές της επιθυμίες και να πει ότι να συντάξουμε μια κοινή επιτροπή, η Επιτροπή Μεταφορών για τις Μεταφορές, ε, η Επιτροπή Βιομηχανίας για την ε, εξόριξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και του καθεξής, ο καθένας με τον πόνο του. Αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε εδώ για ολοκληρωμένη προσέγγιση, πράγμα που σημαίνει σημαίνει ότι δεν πρέπει να κατευθυνθούμε προς μία ή άλλη κατεύθυνση. Θα προτιμούσα ξεχωριστά ε, έγγραφα πολιτικής ε, για την, πολιτική κάθε, για την κάθε πολιτική χωριστά ε, για την Αρκτική. Εδώ όμως θέλουμε ισότιμα να αντιπροσωπευτούν όλες οι πολιτικές, γιατί έτσι πρέπει. Σε σχέση τώρα με τις ε, χώρες της, ε, της δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε αιτήματα και προσδοκίες, λες και ήταν δική μας Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Αν δούμε τον ωκεανό της Αρκτικής, δεν υπάρχει καμία επικράτεια που να, ανήκει, ε, που να ανήκει στην Ένωση. Έχουμε κάποια κράτη-μέλη, εντάξει, αυτό είναι ευπρόσδεκτο, κάποια κράτη-μέλη που είναι πιο δραστήρια, αλλά θα πρέπει τις πολιτικές μας να τις, να τις, ε, ε, να ενεργοποιήσουμε, να ενθαρρύνουμε δηλαδή τα μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου, που είναι και μέλη της Ένωσης, να ε, δράσουν και να προσφέρουμε στα μέλη του Συμβουλίου της Αρκτικής την καλή μας συνεργασία και την πυρογνωμοσύνη που μπορεί ενδεχομένως να έχουμε ως ad hoc παρατηρητές, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το καθεστώς μας, αλλά θα πρέπει να περιοριστούμε και γιατί όπως είπα δεν είμαστε ιδιοκτήτες της Αρκτικής, ωστόσο έχουμε θεμητά συμφέροντα για την ειρηνική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και για την βιώσιμη διαχείριση της περιοχής καθώς και την προστασία των πόρων. Όπως είπα νωρίτερα, βλέπουμε και ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την περιοχή ως μια ειρηνική περιοχή που οι συγκρούσεις που έχουμε με τη Ρωσία και άλλους για άλλες περιοχές δεν θα μας ε, έρθουν ως έκπληξη αλλά θα διατηρήσουμε μια συνεργασία όπου αυτό είναι δυνατόν Ε, συνεργασία με τη Ρωσία ε, για την ε, θάλασσα Μπάρεντς, για τα στόκ, τα αλληλευτικά στόκ, όπου έχουν υποδειγματική συμπεριφορά οι Ρώσοι και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να δείξουμε ότι ακόμα και όταν έχουμε να κάνουμε μια αυταρχική χώρα, αυταρχική χώρα μπορούμε να συνεργαστούμε σε διάφορους τομείς πολιτικής. Θέλουμε να τονίσουμε τα διάφορα κοινά στοιχεία και τις ε, δυνατικές ε, νέε πρωτοβουλίες. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσουν από κοινού την πρόταση για δημιουργία ενός, ε, ομάδα εργασία για τα αρκτικά ζητήματα και μια αντιπροσωπεία για την συνεργασία, τη Βόρεια και την συνεργασία με τις χώρες της Αρκτικής. Αυτό θα ήθελα και εγώ να το ενθαρρύνω, γιατί αυτό θα προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της περιφέρειας αυτής Για την ώρα λοιπόν ως ad παρατηρητές μπορούμε να κάνουμε το ίδιο, δηλαδή να προσφέρουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας. Τουλάχιστον το 2020 να πούμε ότι έχουμε, μάλλον μέχρι το 2020, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με το Συμβούλιο της Αρκτικής, να ενισχύσουμε τους κανόνες ώστε να μην υπάρξουν συγκρούσεις για τους πόρους. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Τώρα για τη συμβιβαστική 2. Ε, θα ήθελα να δούμε αυτές οι γραμμές ε, στις εντός παρανθέσεων να μην περιλαμβάνονται στο τελικό κείμενο ε, και δεδομένης του, του διεθνούς πλαισίου να υπάρξει και μια μεταφορά βιώσιμων ε, προγραμμάτων. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε τον περιορισμό της ανθρώπινης δραστηριότητας σε καθαρά επιστημονικούς στόχους στη συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής. Η παράγραφο, μάλλον το εδάφιο 3 της παραγράφου 6 δεν ζητά αρκετά, γιατί δεν έχει αποδειχθεί η ανεπάρκεια των υποχρεώσεων ε, ε, περιβαλλοντικής αξιολόγησης που ισχύει ήδη για τις χώρες που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Αρκτικής. Το σχέδιο συμβιβαστικής 6 της παραγράφους 13 και 14 δεν θα έπρεπε να είναι ουσιαστικό κομμάτι του κειμένου. Για, κατά τη γνώμη μου που είμαι μέλος της Επιτροπής Αφέτες, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Λίζα Γιακονσάρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές, τον Ούρμαν Σπάιτ και τη Σύρπα Πιετικάινεν, για την πολύ θετική συνεργασία που είχαμε. Αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα καθ' όλη την επεξεργασία της έκθεσης αυτής ήταν να γνωρίσουμε το έργο που έχει επιτελέσει το Αρκτικό Συμβούλιο. Και ας έχουμε κατά νου ότι θα πρέπει αυτό να φαίνεται κάπου και στο ίδιο το ύφος της έκθεσης. Μια έκθεση η οποία ακόμα βρίσκεται σε φάση εκπόμνησης, μην το ξεχνάμε. Ουσιαστικά συμφωνώ με τους προορίσαντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά εμφανίζεται υπεροπτική. Μια να λειτουργεί λίγο σαν μεγάλο αδερφό απέναντι σε χώρε οι οποίε βρίσκονται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια λοιπόν τη πολιτική για την Αρκτική είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τη θετική συνεργασία που θα πρέπει να έχουμε με χώρε όπω ο Καναδά, η Ρωσία, η Ισλανδία, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώ το λόγο δεν θα πρέπει εμεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιτάσσουμε στι άλλε χώρε τι ακριβώ θα πρέπει να κάνουν και μάλιστα αφιψηλού. Νομίζω ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε στα πλαίσια μιας επικοδομητικής συνεργασίας. Και κάτι ακόμα. Στην έκθεση αυτή προσθέσαμε και την βόρεια διάσταση, την εταιρική σχέση της βόρειας διάστασης. Ξέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ωστόσο όμως είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, ιδιαίτερα ρεαλιστικό. Έχει ως στόχο να καταλήξει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχει να κάνει με τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ρωσίας, της Ιρλανδίας και του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε περισσότερο στους στόχους της ε, βόρειας διάστασης. Ο Καναδά και οι ΗΠΑ έχουν ακόμα το καθεστώ του παρατηρητή στα πλαίσια τη βόρεια διάσταση. Θα πρέπει λοιπόν κάπου στο κείμενο να γίνεται και μία μνήα στο πρόγραμμα αυτό. Επίση, έχουμε συζητήσει πάρα πολύ το ζήτημα τη Ρωσία και με αφορμή την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι πολλές φορές η προσέγγιση μας, ιδίω στην έκθεση αυτή, είναι θετική και θα πρέπει να είναι θετική, ιδίω σε ένα πλαίσιο όλο και αυξανόμενων εντάσεων. Πρέπει να κάνουμε κάθε το δυνατό προκειμένου να διασφαλίσουμε μια θετική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, ιδίω σε τομείς που η συνεργασία αυτή έχει ήδη αποβεί θετική στο παρελθόν. Και αναφέρομαι εδώ πέρα στη μνήμα που γίνεται όσον αφορά την στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας στην περιοχή της Αρκτικής. Ένα, ένα από τα δυνατά σημεία της έκθεσης έχει ήδη αναφερθεί από τους προαλήσαντες, το ότι δηλαδή η έκθεση αυτή όλο και περισσότερο πλέον τονίζει την ανάγκη συμπερίληψης των αυτόχθονων και τοπικών πληθυσμών στη λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι πληθυσμοί αυτοί όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την περιοχή τους. Νομίζω ότι ο φιλόδοξος αυτός στόχος είναι πάρα πολύ σημαντικός, καθότι μιλάμε για την πρώτη γενιά πλέον αυτόχνων πληθυσμών που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην εκπόνηση και το σχεδιασμό της στρατηγικής για την Αρκτική. Είναι επίσης πολύ σημαντικό, πέρα από την κοινοτική χρηματοδότηση, πέρα από τα κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, να κινητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης της πολιτικής ε, για την Αρκτική. Να καταφέρουμε δηλαδή να δώσουμε ακόμα και στη χρηματοδότηση μια πιο διεθνή διάσταση. Να καταφέρουμε να έχουμε ακόμα και έργα για την κατασκευή υποδομών. Και επίσης, ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ευθύνη των ε, πληθυσμών της Αρκτικής η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τι κλιματικέ αλλαγέ. Δεν θα πρέπει εμεί να λαμβάνουμε αποφάσει που τελικά τιμωρούν του πληθυσμού αυτού, που ε, δεν είναι καθόλου υπεύθυνοι για την υφιστάμενη κατάσταση. Ανταυτού νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε μέτρα μετριασμού των κλιματικών αλλαγών και μέτρα τα οποία θα πρέπει να συνδυαστούν με οικονομικά μέτρα και με άλλα εργαλεία τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την επιτόπου κατάσταση. αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την εργασία που γίνεται στα πλαίσια του Αρκτικού Συμβουλίου. Ιδίω την εργασία που κάνει το Αρκτικό Συμβούλιο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκεκριμένων προγραμμάτων. Και επαναλαμβάνω ότι δεν θα πρέπει εμείς να επιβάλλουμε συγκεκριμένε πολιτικές ιδίω όσον αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, σε άλλε χώρε του Αρκτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι επί ίση όρη θα πρέπει να συνεργαστούμε ακόμα και για τα περιβαλλοντικά ζητήματα με τι χώρε αυτέ. Του των εκθέντων, χαίρομαι πάρα πολύ που οι συνάδελφοι οι συνεισηγητέ αποδέχθηκαν και την ιδέα τη κοινωνική ευθύνη, μια κοινωνική εταιρική ευθύνη για την περιοχή τη Αρκτική. Εταιρική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά δηλαδή τι επιχειρήσει εκείνε οι οποίε δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή της Αρκτικής. Και επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπω είπα πριν από λίγο, να έχουμε και την απαραίτητη υποδομή στην περιοχή αυτή, στην οποία θα βασιστούν και μελλοντικέ οικονομικέ δραστηριότητε. Αναφέρομαι εδώ πέρα τόσο στι παραδοσιακέ μορφέ υποδομών, όσο και στι νέε ψηφιακέ ή ασύρματε συνδέσει που θα πρέπει να πτυχθούν περισσότερο στην ελόγω περιοχή. Τέτοια προγράμματα, τέτοια έργα πιστεύω ότι θα πρέπει να τα υποστηρίξουμε. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην περιοχή τη Τρακτική για τι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι εμεί ω Ευρωβουλευτέ το είχαμε προτείνει αυτό ήδη από πέρυσι. Είναι λοιπόν πάρα πολύ θετικό που έχουμε και την υποστήριξη πλέον των ίδιων των βουλευτών των εθνικών βουλευτών από τις περιοχές της Αρκτικής, από τα κράτη-μέλη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στην περιοχή της Αρκτικής. Υπάρχει μια σύμπνοια μεταξύ Ευρωβουλευτών και Εθνικών Βουλευτών όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι εκκρεμούν ακόμα δύο-τρει συμβαστικέ τροπολογίε, επί των οποίων δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα επίσημα. Είμαι σίγουρο όμω ότι θα το πετύχουμε και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Ντόρμαν έχει τώρα το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ και θα μιλήσω δανέζικα, στη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές που κατέρτισαν την έκθεση αυτή. Και όπως γνωρίζετε, βασικά οι αρκτικές ε, χώρες, οι χώρες της Αρκτικής και οι κυβερνήσεις τους είναι αυτές που καθορίζουν την πολιτική για την Αρκτική. Σε κάποιους τομείς ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει και καταβάλλει κοινέ προσπάθειες, ε, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την κλιματική πολιτική, την πολιτική για το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το μεγαλύτερο χορηγό και το μεγαλύτερο παράγοντα, αν θέλετε, ε, στην πολιτική για την Αρκτική μέσω από το πρόγραμμα πλαίσιο 6 και 7. Έχουμε 200 εκατομμύρια τα οποία έχουμε ορίσει για το 2020. Εδώ έχουμε προβλέψει και επιπλέον ε, πόρου και κονδύλια. Παίζει λοιπόν σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να επικεντρωθώ στι σχέσει μα με τη Ρωσία. Αληθεύει όντω ότι η Ρωσία αυξάνει διαρκώ την στρατιωτική της παρουσία στην ε, περιοχή της Αρκτική και εξοπλίζεται. Παρ' όλα αυτά είναι απαραίτητο να διατηρηθούν καλά σχέσει με τη Ρωσία. Αν ε, οι χώρε τη Αρκτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να αντιμετωπίσουν τι βασικέ προκλήσει και να υπάρξει και μια διεθνή σύμβαση για την Αρκτική, θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τι ε, συνομιλίε με τη Ρωσία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την Ρωσία στην Αρκτική, στην, σε ό,τι αφορά την βόρεια διάσταση. Και έχω συνομιλήσει με τη Ρωσία σε διάφορες περιστάσεις και η Ρωσία αντιλαμβάνεται τη σημασία της αρκτικής συνεργασίας. Αν θέλουμε να έχουμε μόνιμη θέση, μόνιμη παρατροπή στο Συμβούλιο της Αρκτικής, θα πρέπει να διατηρήσουμε μία αλφα σχέση με την ε, Ρωσία. Και να σας πω και από το Δανέζικο Τμήμα του Στρατού που ασχολείται με τις θαλάσσιες διασώσεις, η συνεργασία με τη Ρωσία είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την Αρκτική, γιατί υπάρχει η συνεργασία και με την Βερλανδία. Ε, Έχουμε βουλευτές ε, από τη Βερλανδία στο Δανέζικο Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο λόγια παραπάνω. Για τις διαπραγματεύσεις με, το... με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά την Αρκτική. Ωστόσο, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν και για τους αυτόχθονες σε ό,τι αφορά και τα τοπικά προϊόντα και όχι να αντιμετωπίζουμε την Αρκτική ως μια περιοχή όπου δεν συμβαίνει τίποτα. Η ε, κυρία Νταλή, σας ευχαριστώ. Εκπροσωπώ την κυρία Σαλτεμόζε και θα ήθελα εξ ονόματός της να ευχαριστήσω καταρχάς τους δύο συνεισηγητές. Επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους κοιοδές για τη συνεργασία τους για το θέμα αυτό. Είμαστε ικανοποιημένοι με τις ε, συμβαστικές προτάσεις και είμαστε βέβαιοι ότι αν συνεχίσουμε με τον τρόπο αυτό θα βρούμε και περαιτέρω συμβαστικές λύσεις από πλευράς ε, ε, σοσιαλιστών και δημοκρατών και σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος θέλουμε να υπάρχει μεν και περιβαλλοντική προστασία υψηλής ποιότητας, αλλά να γίνονται σεβαστές και οι ανάγκες των λαών και των κυβερνήσεων στην Αρκτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς θα πρέπει να συμβάλλει στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη της Αρκτικής, αλλά παράλληλα είναι σημαντικό αυτό να συνάδει και με τις επιθυμίες των λαών της Αρκτικής. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η εξέλιξη θα λάβει υπόψη ακριβώς και τους αυτόχθονες στην Αρκτική και ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις δυνατότητες οικονομικής τους ανάπτυξη θα πρέπει να έχουμε διαρκώ υπόψη ότι η Αρκτική, σε αντίθεση με την Ανταρκτική, είναι μια περιοχή που κατοικείται. Και το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής είναι υπό εθνική δικαιοδοσία. Αυτό τι σημαίνει, ότι αυτές οι χώρες, αυτοί οι λαοί θα πρέπει να αποφασίζουν για την νομοθεσία και οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιβληθεί στην περιοχή. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη μελετών αντικτύπου. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει τι χώρε αυτέ προ την κατεύθυνση αυτή. Α, παρ' όλα αυτά όμω, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε να είναι υποχρεωτική υποβολή τέτοιων μελετών αντικτύπου στην Αρκτική. Και εξ ονόματος λοιπόν της Κριστέλ θα ήθελα να πω ότι η έκθεση μας φαίνεται ισορροπημένη. Σας ευχαριστούμε και προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία για να ρυθμίσουμε και τα εκκρεμή ζητήματα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ λέει και πρόεδρος η κυρία Γιατενμάκη. Ευχαριστώ. Να πω και δύο λόγια για την γεωγραφική κατάσταση και τη διεθνή συνεργασία. Νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι και μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι σε ό,τι αφορά την περιοχή της Αρκτικής. Δεν υπάρχουν τρυφές και εντάσεις. Μην σας πω ότι είναι η μοναδική περιοχή στη γειτονιά μας. Όπου υπάρχει μια τακτική συνεργασία και όλοι στις συναντήσεις ε, του Συμβουλίου Αρκτικής και άλλε συναντήσει μεταξύ των κρατών μελών δηλώνουν ότι η συνεργασία πραγματικά είναι εξαιρετική. Άρα πιστεύω ότι σκοπός μας θα πρέπει να είναι και στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχιστεί η καλή συνεργασία Τώρα που μάλιστα όλος ο υπόλοιπος κόσμο μαστίζεται από εντάσει και τριβέ, αυτό πραγματικά είναι κάτι το ασυνήθιστο και θα πρέπει να διατηρηθεί θυσία. Να πω τώρα δύο λόγια για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την ε, περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά την Αρκτική. Πιστεύω ότι αυτά είναι βασικά ζητήματα στην έκθεση. και εγώ και η ομάδα μου υποστηρίζουμε την παράγραφο 6. Είμαι πεπισμένη ότι θα βρούμε μια τύπωση που θα τη χάνει τις υποστηρίξεις της πλειοψηφίας της Επιτροπής, γιατί, όπως σας είπα, αυτό αποτελεί από τα βασικά ζητήματα. Τώρα, να εκφράσω και κάποιες επιφυλάξεις ότι αφορά την παράγραφο 7 όπου αναφέρεται η επιτυχής εφαρμογή της μελεπισταντικ ω ως προδιαγραφή, ως όρος. σε ό,τι αφορά την πολιτική για την Αρκτική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα τι Αυτό συνάδει με τους κανόνες της ενίας αγοράς. Μα ούτε για το σκοπό αυτό είναι ωφέλιμη και χρήσιμη η προδιαγραφή αυτή. Είμαι βέβαιη ότι μπορούν να έρθουν μεγάλες επιχειρήσεις από την εκτός Αρκτικής και να πολλούν τα προϊόντα τους. Και τελικά ο κόσμος ο οποίος ζει εκεί, που δεν έχει μεγάλες επιχειρήσεις, δεν έχει πόρους για να κάνει τέτοιες μελέτες αντικτύπου ή να τις ε, αναθέσει σε κάποια εξωτερική εταιρεία, τελικά αυτοί τα είναι που θα ζημιωθούν. Είναι δυνατόν αυτός να είναι ο σκοπός που επιδιώκουμε. Εν πάση να ευχαριστήσω τους εισηγητές και όσους συνεργάστηκαν μαζί μας και πιστεύω ότι θα πετύχουμε σε τελική ανάλυση πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος ε, της συναδέλφου Φωτίγα, που είναι ε, η σκιώδηση εισηγήτριά μας για την Ισιάρκεια που δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ, αλλά και προσωπικό, θα ήθελα να σας διαβιβάσω τα σχόλιά μας σε σχέση με το σχέδιο κειμένου. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τους συνεισηγητές που προετοίμασαν ένα περίπλοκο αλλά όχι και τόσο τεχνική έκθεση περίπλοκη αλλά όχι και τόσο τεχνική που συνδυάζει τα πολιτικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι δύο πτυχέ είναι πολύ σημαντικέ ε, για την Αρκτική και το κείμενο αντικατοπτρίζει αυτή την δύσκολη ισορροπία. Η πρώτη πτυχή, κατά την άποψή μα και κατά την άποψη των μονομένων ε, ε, κρατών μελών, αποτελεί μια σημαντική συμβουλή, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ερευνητικά κέντρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστούν και να προχωρήσουν εργασίες σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει δεν να συντονιστούν ακόμη καλύτερα αυτές οι προσπάθειες ε, και μάλιστα να οδηγήσουν σε αύξηση της χρηματοδότησης από πλευράς της Ευρώπης κατά την απόψή μας. Επίσης, όλο ένα και μεγαλύτερη είναι η γεωπολιτική σημασία της περιφέρειας ε, αυτής και Οποιοδήποτε γεγονός στην Αρκτική έχει αντίκτυπο και στις υπόλοιπες περιφέρειες του κόσμου. Ένα αρνητικό σημείο σε μήνυμα είναι η ανεπαρκής προσοχή που δίνεται στο ρόλο των δυνητικά αποστοθεροποιητικών της Ρωσίας, κυρίως ενώπιον της μαζικής ανάπτυξης των στρατιωτικών υποδομών, αλλά και της ολοένα μεγαλύτερης παρουσίας του στρατού στην περιοχή. Συμβιβαστική 4 γίνεται λόγος για το φόρμα Τη της για να περιγραφεί ο διάλογος ανάμεσα στους παρατηρητές και τη ο Συμβούλιο της Η, Το ECR θα ήθελε να υπάρξει αυτή η αναφορά στη Συμβαστική 4 γιατί έτσι καθορίζεται καλύτερα αυτή η διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Λόζινγκ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τους συνεισηγητές. Ήταν φαντική και επικοδομητική η συνεργασία σας. Ευχαριστώ. Και εγώ και η ομάδα μου ε, με θετικό μάτι βλέπουμε την έκθεση σε μεγαλύτερο βαθμό. Και θεωρώ ότι και η συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος ήταν παρακολουθητική. Κάτι άλλο που είναι επίσης ε, σημαντικό είναι να συνεχίσει να είναι μεγάλη η συνεργασία και η συμπερίληψη των ε, αυτόχθονων πληθυσμών σε ό,τι αφορά την οικονομική, πολιτική ανάπτυξη την, ε, και όλα τα στοιχεία τα οποία ανέφεραν και οι συνάδελφοι προηγουμένω, περιβαλλοντική προστασία και το καθεξής. Τώρα, Ένα σημαντικό θέμα είναι η προστασία του ευαίσθητου περιβάλλοντος. Και υπάρχουν σημαντικά στοιχεία τα οποία και στο μέλλον θα συνεχίσουν να διδραματίσουν σημαντικό ρόλο και πολλές από τις τροπολογίες ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Το σχέδιο τονίζει ότι μια συμφωνία θα πρέπει να επιτευχθεί μια κοινή συμφωνία για την Αρκτική, η οποία θα αποτελέσει ένα κοινό κληροδότημα και ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για ε, ελληνικού ε, σκοπούς ανάπτυξης. Και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνθήκη η οποία θα προσωμιάζει στη συνθήκη που υπάρχει για την αντακτική, που δημιουργεί, αν θέλετε, ένα πλαίσιο για μια ειρηνική συνεργασία χωρίς ριβές, χωρίς ε, προστριβές, χωρίς ζητήματα μεταξύ των κρατών εθνών. Και επίσης καλυσορίζουμε το γεγονός ότι η έκθεση ε, τονίζει την ε, αποτροπή στρατιωτικοποίηση της περιοχής. Και εδώ θεωρούμε ότι θα μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παραμείνει η περιοχή ως μια περιοχή χαμηλών ε, εντάσεων. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι η... παρουσιάζεται με κάπως μονομερή τρόπο η επικέντρωση στα θέματα της αρκτικοποίησης της Αρκτικής. Στο πλαίσιο όμως αυτό, αυτό που είναι σημαντικό είναι να κοιτάξουμε την γενικότερη στρατικοποίηση της περιοχής της Αρκτικής από τη Ρωσία και από τον ΝΑΤΟ, την ΣΥΠΑ, τον Καναδά, τη Δανία, την Νορβηγία. Αυτά όλα πρέπει να τα αναφέρουμε. Ας θυμηθούμε την ε, πρωτοβουλία Arctic Challenge σε ό,τι αφορά τον αέριο χώρο του ΝΑΤΟ το 2015. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν για την αύξηση των καναδικών αεροσκαφών δεν συνέβαλε σε καμία περίπτωση στην περαιτέρω κατανόηση και στην εμβάθυνση της εργασίας στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Μάισνερ τώρα. Σα ευχαριστώ. Θα μιλήσω και εγώ στα γερμανικά, μια και μιλήσει και προλαλήσασα. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλου όσοι συνεργάστηκαν για την έκθεση αυτή και θα ήθελα να κάνω μόνο μια σύντομη προσθήκη, αν μου επιτρέπετε. Είπε προηγουμένω ο κ. Γκάλαρο ότι σχεδόν όλε οι επιτροπέ συνεργάστηκαν για την έκθεση αυτή. Όντω, είναι κάρσιο το ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να υπογραμμίσω και κάτι άλλο το οποίο δεν αναφέρθηκε σήμερα είναι και αυτή η ενσωματωμένη πολιτική για τις θάλασσες, η οποία τι λέει, ότι πρόκειται για μια περιοχή η οποία περιλαμβάνει πολύ πιο πολλά από θαλάσσια από θαλάσσια Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι και να ληφθούν υπόψη όλα αυτά τα συμφέροντα. Και φυσικά αυτό συμπεριλαμβάνει και τα συμφέροντα του περιβάλλοντος, των χώριων πληθυσμών, τα οικονομικά συμφέροντα και θέματα άμυνας, προφανώς. Αυτό Λοιπόν, το υπογραμμίζω γιατί αυτή η προσέγγιση η οποία έχει σχεδόν κλείσει τη δεκαετία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντική και θεωρείται δεδομένη ocean governance για κυβέρνηση διαχείριση των ωκεανών. Αυτό το συζητάμε, αυτό σχετίζεται με την έκθεση. Αλλά έχω γενικά την εντύπωση ότι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον υπόλοιπο κόσμο όλο και πιο πολύ και πιο μεγάλο ρόλο παίζουν οι θάλασσες. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπήρχε μία επιτροπή η οποία θα ασχολείται με θέματα θάλασσας. Ίσως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε και την ονομασία της Επιτροπής Αλίας. Ξέρω ότι συμφωνεί και ο Επίτροπος, ο αρμόδιος με το θέμα αυτό. Θα ήταν καλό λοιπόν να ληφθούν αυτά υπόψη με ένα συνολικό στον τρόπο. Και φυσικά εν γέννη η Αρκτική είναι σημαντική για μας και για λόγους ε, οικονομικούς αλλά και για λόγους άμυνας αλλά να μην ξεχνάμε και τη σημασία της προστασίας της φύσης. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις νέες αυτές τις ζώνες. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά και εγώ να ευχαριστήσω του δύο εισηγητέ. Νομίζω ότι συνεργαστήκαμε πολύ θετικά. Και νομίζω ότι όλοι εκτελήθηκαν σε ένα πολύ θετικό πνεύμα συνεργασία μεταξύ σκιωδών εισηγητών και συνεισηγητών. Ο κύριο Γκάλερ είπε ότι δεν μιλάμε εδώ πέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υποτίθεται ότι δεν δραματίζει συγκεκριμένο ρόλο στην περιοχή. Εν μέρει αυτό ισχύει. Αλλά δεν μιλάμε εδώ πέρα μόνο για την περιοχή της Αρκτικής μεμονωμένα. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε στη σημερινή εποχή και μιλάμε για και πολύ σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Η κλιματική αλλαγή είναι μία πρόκληση, παγκόσμια πρόκληση και αν δεν ασχοληθούμε με το μετριασμό τη, αν δεν ασχοληθούμε με την αντιμετώπιση τη, τότε θα αντιμετωπίσουμε δεινέ επιπτώσεις στο μέλλον. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να πληγούν πάρα πολλοί άνθρωποι, εκατομμύρια ανθρώπων στον Παγκλατέ, σε νησιωτικά κράτη. Η ίδια η κατάσταση της ε, νεκρής θάλασσας ε, κινδυνεύει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα κοινό όραμα για το μέλλον. Και α μην ξεχνάμε ότι έχουμε και κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται στην περιοχή τη Αρκτική. Γι' αυτό και μόνο το λόγο πρέπει κι εμεί να έχουμε μια κοινοτική πολιτική για την Αρκτική. Το κοινικό στην όλη υπόθεση είναι ότι όσο περισσότερο λιώνουν οι πάγοι στην περιοχή, τόσο αυξάνονται οι ευκαιρίε εξόριξη φυσικού αερίου και πετρελαίου σε περιοχέ που ήταν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο εξαιτία των παγατώνων στο παρελθόν και όσο περισσότερο εκμεταλλευόμαστε τους σπόρους αυτούς, τόσα περισσότερα προβλήματα κλιματικά δημιουργούμε και τόσα περισσότερα παγκόσμια προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Είναι αρκετά ηρωνικό αυτό. Ας δούμε λίγο τα αριθμητικά δεδομένα, τα οποία δεν τα είχαμε στην αρχή της ε, έκθεσης. Αν δούμε κάποια στατιστικά αριθμητικά δεδομένα, βλέπουμε ότι εν μέσω του χειμώνα η θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί υψηλότερη από ό,τι λογικά θα ήταν αυτή την εποχή στην περιοχή της Αρκτικής και καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί μια καταστροφική εξέλιξη για την περιοχή. Θα πρέπει επίσης να δούμε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα αρκτικά χωρικά ύδατα και την ίδια την Αρκτική. Όσοι προερχόμαστε από αρκτικά κράτη-μέλη, έχουμε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να εξηγήσουμε στους υπόλοιπους ότι ένα μεγάλο μέρος της Βόρειας Σουηδίας, για παράδειγμα, εντάσσεται στην αρκτική περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάπως προβληματικό κάθε φορά που μιλάμε για προστασία της Αρκτικής. Γιατί από σημασιολογικής πλευράς ουσιαστικά αναφερόμαστε και σε κάποια τμήματα της Σουηδίας, όπου ζουν κανονικοί κάτοικοι και όχι μόνο αυτόχθονες, όλοι μας ζούμε στην περιοχή αυτή και όλοι θέλουμε να έχουμε σιδετρομικές υποδομές ή και άλλες υποδομές οι οποίες να λειτουργούν φυσιολογικά. Υπάρχουν λοιπόν πολλές περιοχές αρκτικής οι οποίες ε, κατοικούνται κανονικά και όχι μόνο από αυτόχθονες πληθυσμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω να προστατεύσουμε και τα ύδατα των περιοχών αυτών, ιδίω περιοχές περιοχέ εκείνε που έχουμε σημαντική τήξη των παγετώνων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιε προστατευόμενες περιοχές ή σε ένα μορατόριο τουλάχιστον ...στην αφορά την εκμετάλλευση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ένα καθοριστικό στοιχείο στρατηγική αυτή θα πρέπει να είναι η διασύνδεση της στρατηγική αυτής με την πολιτική μας για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και να συνδεθεί επίση και με τι αρνητικέ επιπτώσει που έχει η εξόριξη πετρελαίου, επιπτώσεις οι οποίες αφορούν το σύνολο του πλανήτη όπως σας είπα. Πολλοί αναφέρθηκαν στο σημείο 6 της έκθεσης που είχε να κάνει με την εξολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της έκθεσης αυτής, ε, όχι το πιο σημαντικό αναγκαστικά, αλλά ένα από τα πιο καθοριστικά σημεία αυτής της έκθεσης. Νομίζω λοιπόν ότι ε, σε βάθος χρόνου θα πρέπει αυτή η αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων να γίνει δεσμευτική και υποχρεωτική. Ουσιαστικά καλούμε τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο Αρκτικό Συμβούλιο να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα. Καταλαβαίνω αυτό που λένε οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Όντως, το σύνολο της περιοχής Αρκτικής δεν είναι το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο ευάλωτο, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Οι νότιες κυρίως περιοχές της Αρκτικής ενδεχομένως να μην πλήττονται τόσο πολύ από τα καιρικά φαινόμενα όσο οι πιο ευάλωτες βόρειες περιοχές, οι περιοχές οι οποίες έχουμε κυρίως ύδατα και παγετώνες. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά το σημείο 7. Ήδη στις πιο ευάλωτες αυτές περιοχές κάνουμε αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου για όλα τα προγράμματα τα οποία ενδεχομένως να έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε και στο μέλλον. Αυτό άλλωστε επιβάλλουν οι ίδιοι οι ενωσιακοί κανόνες που υφίστανται αυτή τη στιγμή. Θεωρώ λοιπόν ότι το σημείο 6 είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γενικότερο ζήτημα που έχει να κάνει με την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι καθοριστικό και θα πρέπει η αξιολόγηση αυτή να είναι υποχρεωτική και δεσμευτική. Θα ήθελα να προωθήσω περισσότερο το σημείο αυτό. Δυστυχώ γνωρίζω δεν υπάρχει πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτού. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά του εισηγητέ και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα αναπομείνητα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, λέει ο Πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ενδεχομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να θέλουν να πάρουν τώρα το λόγο. Ο κύριο Ντεπιέγα από την DG Mare. Ενδεχομένω θέλετε να προσθέσετε κάτι εσεί. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε σήμερα ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας την κοινή αυτή δήλωση, την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά την ολοκληρωμένη στρατηγική για την Αρκτική. Η ίδια Αρκτική είναι μια ολοκληρωμένη σφαιρική περιοχή τουλάχιστον στην αντιμετώπιση που χαίρει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθότι κινητοποιούνται πολλέ διευθύνσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ίδια η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση, αλλά εδώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπω ότι συνεργάζονται δύο τουλάχιστον επιτροπέ. Καλωσορίζουμε λοιπόν το σχέδιο έκθεση των δύο επιτροπών σα, που στηρίζουν ουσιαστικά την κοινή μα δήλωση και στηρίζουμε επίσης και τις γνωμοδοτήσεις άλλων επιτροπών που τονίζουν πάρα πολύ τα ζητήματα λίας και τα ζητήματα εμπορίου. Καλωσορίσουμε επίσης την υποστήριξη των δύο συνεισηγητών, καθώς επίσης και των υπολείπων ευρωβουλευτών από διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κοινή αυτή λοιπόν δήλωση βασίζεται σε μια πρώτερη πρωτοβουλία και βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη πολιτική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αλλά και των ευκαιριών στην περιοχή της Αρκτική και για να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την ήδη σημαντική παρουσία μας στην περιοχή αυτή. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο ρυθμιστικό πλαίσιο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αρκτική συνδέονται άρρηκτα. Οι επιπτώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αρκτική αλλά και τη Αρκτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθίστανται όλο και πιο σημαντικέ και όλο και πιο σαφεί. Και στο περιβάλλον αυτό μπορούμε να εντάξουμε και τα σχόλια τη κυρία Γιατανσάρη, το ότι όντω έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία στα πλαίσια του Φόρουμ τη Βόρεια Διάσταση. Η Αρκτική λοιπόν όλο και περισσότερο συμβάλλει στι πολιτικέ για την κλιματική αλλαγή και βλέπουμε ότι ω περιοχή υπερθερμαίνεται με διπλάσιου ρυθμού σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη και το αρκτικό αυτό περιβάλλον τροποποιείται, πράγμα το οποίο τροποποιεί επίσης και τις συνθήκες διαβίωσης για τη χλωρίδα και την πανίδα. Παγκόσμιε όμω είναι και επιπτώσει στα γενικότερα πρότυπα κλιματολογικά και μετεωρολογικά τα οποία εμφανίζονται παγκοσμίω και που συμβάλλουν σε αύξηση τη στάθμη τη θάλασσα. Επίση βλέπουμε ότι ε, λόγω της ε, τήξη των μόνιμων των αυξάνονται και εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο απαιτείται κοινή συνεργασία ιδίω στον τομέα τη επιστημονική έρευνα. Οι προκλήσεις σε μια τέτοια κλίμακα είναι πάρα πολύ σημαντικέ και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από μια χώρα μόνη τη. Επιβάλλεται λοιπόν διεθνή συνεργασία και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να καταλάβουμε καλύτερα πώ λειτουργούν οι όλε αυτέ μετρολογικέ διαδικασίε και ποιε είναι οι επιπτώσει που θα έχουν. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η διεθνή επιστημονική συνεργασία στην Αρκτική μέσω των προτάσεων που γίνονται και στην κοινή δήλωση και μέσω και των πολύ θετικών προτάσεων που έκαναν ορισμένοι ευρωβουλευτέ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υποστήριξη. Θέλουμε και βιώσιμη ανάπτυξη για τους ε, τοπικούς πληθυσμούς της Αρκτικής. Η Αρκτική όπως είπατε και εσείς στις παρεμβάσεις σας, απαριθμεί 4 εκατομμύρια κατοίκους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις χρηματοδοτήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή αυτή, δίνοντας προτεραιότητα στην γαλάζια και πράσινη ανάπτυξη. Μπορεί όντω να προωθήσουμε και την καινοτομία και την ευφυή ανάπτυξη στην περιοχή αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει του αυτόχθονε πληθυσμού να χρησιμοποιήσουν το δυναμικό του με τον ευφιέστατο δυνατό τρόπο και να ευχαριστήσω εδώ πέρα και τον κύριο Ντόρμαν ο οποίος είπε ότι οι πρωτοβουλίες που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ως στόχο την ισορροπημένη ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού των ατόπων της περιοχής αυτής και όχι μόνο την εκμετάλλευση των εθνικών πόρων. Το σχέδιο λοιπόν έκθεσης πολύ σωστά τονίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να λάβει χώρα μόνο αν οι επιπτώσεις, οι επιπτώσεις των προγραμμάτων αυτών ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Αρκτικό Συμβούλιο, ιδίως όσον αφορά την, τον στο χαρακτήρα της περιοχής αυτής σε νοσιακό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξολογίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα μέσα αυτά, τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται και στην περιοχή της τρακτικής. Αν τα εφιστάμενα λοιπόν αυτά εργαλεία χρησιμοποιηθούν πλήρως, τότε έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε στην περιοχή αυτή όντως προστατεύουν το περιβάλλον και όντως είναι βιώσιμα. Η πρόοδος που έχει ήδη σημειωθεί στην εφαρμογή της κοινή δήλωσης θα πρέπει να αναφερθεί. Θα πρέπει σήμερα να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της ανακοίνωσή μας ιδίως όσον αφορά την δημιουργία ενός προσωρινού φόρουμ των εμπλεκόμενων μερών, όπου συμμετέχουν οι αυτόχθονες, οι κυβερνήσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να γίνει η ιεράρχηση επενδυτικών προτεραιοτήτων για τα επόμενα χρόνια. Το φόρουμ αυτό έχει ήδη συσταθεί και έχει ήδη συνεδριάσει τρεις φορές. Η επόμενη συνεδρίασή του θα γίνει με την ευκαιρία του Arctic Frontiers Conference στα τέλη Ιανουαρίου. Και η Επίτροπος Βέλε θα είναι παρούσα. Και θα συνεδριάσει το φόρουμ αυτό και τον Ιούνιο στα πλαίσια ενός μιας υψηλόβαθμης εκδήλωσης για την αρκτική πολιτική. Η εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα στη Φιλανδία και θα συμμετάσχει η κυρία Μογκερίνη, η και αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και ο Επίτροπος ε, Θαλασσίων Υποθέσεων και Περιβαλλοντικών Υποθέσεων ΒΕΛΑ. Συνεχίζουμε τη συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τους αυτόχθονους πληθυσμούς. Θέλουμε να έχουμε έναν ετήσιο διάλογο με τους πληθυσμούς αυτούς στα πλαίσια της υψηλόβαθμης αυτής εκδήλωσης που θα λάβει χώρα τον Ιούνιο. Και να πω κάτι και για τη διακυβέρνηση των ωκεανών και για την αλία στην περιοχή της Αρκτικής. Η κοινή αυτή λοιπόν ανακοίνωση για την Αρκτική συνάδει και συνδέεται με την κοινή ανακοίνωσή μας για τη διακυβέρνηση των ωκεανών που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί σήμερα δεν αναγνωρίζουν εθνικά σύνορα, αυτό το ανέφεραν και ορισμένοι ευρωβουλευτέ. Και συμφωνούμε απόλυτα με αυτό. Έχουμε εντοπίσει λοιπόν τρει τομεί προτεραιότητε για ανάληψη δράση. Πρώτον, έγκριση του πλαισίου διακυβέρνηση, διεθνούς πλαισίου διακυβέρνηση για τους ωκεανούς, να καλύψουμε όλα τα κενά και να βελτιώσουμε το στονισμό μεταξύ περιφερειακών, διεθνών και τοπικών οργανισμών, να μειωθεί η αθρική πίεση, ανθρώπινη πίεση στους ωκεανούς και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια γαλάζια οικονομία. Και τρίτον, θα πρέπει να ενισχύσουμε την διεθνή συνεργασία, επιστημονική συνεργασία όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων για του ωκεανού. Όπω σα είπα, πρέπει να καλύψουμε τα φυστάμενα κενά και όπως είπε και ο κύριος Γκάλερ πριν από λίγο, βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια των διαπραγματεύσεων και καταλήξουμε σε μια διεθνή συμφωνία για την αποφυγή της παράτυπης και παράνομης αλίας στην περιοχή της Αρκτικής. Και αν η συμφωνία αυτή εγκριθεί και γίνει δεσμευτική όπως το ελπίζω, θα καλύψει ένα τεράστιο νομικό κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. Εμπλεκόμαστε λοιπόν εμεί σε αυτό, σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω εμπλεκόμαστε και σε άλλε διεθνεί συνεργασίε, οι οποίε λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή για την σύναψη συμφωνιών για του ε, ωκεανού. Όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια του διεθνού δικαίου για τη θάλασσα και με τη συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών. Εν κατακλείδη λοιπόν, η κοινή αυτή δήλωση για την Αρκτική θα δοκιμαστεί ιδίω στην εφαρμογή τη. Η επιτυχία τη ουσιαστικά θα κρυφθεί από την εφαρμογή τη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει την ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, καθώ επίση και με τα εμπλεκόμενα μέρη από το Συμβούλιο τη Αρκτική. Δεν ξέρω αν συναδελφοί μου από τι άλλε διευθύνσει θέλουν ε, να πάρουν και αυτή το λόγο. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό και σε ευχαριστώ για τη γενικότερη υποστήριξή σα. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις Επιτροπές για την πολύ επικοδομητική συζήτηση που είχαμε σήμερα και για την υποστήριξή σας στην κοινή δήλωση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, προκλήσεις ε, ε, ασφάλειας σε αυτή την περιοχή και αντικατοπτρίζονται στην παγκόσμια στρατηγική για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Και νομίζω πως όλοι θέλουμε να διατηρήσουμε την Αρτική ως περιοχή χαμηλών εντάσεων και αυτό σημαίνει επιλεκτική συνεργασία με τη Ρωσία και έχουμε διάφορες, ε, διάφορα φόρα. Το Συμβούλιο της Αρτικής αναφέρθηκε και θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας. για την συμμετοχή της Ένωσης ως παρατηρητής σε αυτό το Συμβούλιο, αλλά υπάρχουν και άλλα φόρα όπως ε, το πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης, επίσης το Συμβούλιο Μπάρεντς Αρκτικής και σε όλα αυτά τα πλαίσια συνεχίζονται οι εργασίε. Βεβαίω έχουμε περιορισμού σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας, αλλά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε κυρίω στο περιφερειακό επίπεδο. Και εδώ θέλω να αναφέρω τα, προγράμματα, τα δυσυνοριακά προγράμματα συνεργασία, που είναι ενεργά και που συμβάλλουν στην υποστήριξη της μεγαλύτερης συνεργασίας στην Αρκτική. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων τη σημερινή. Σας ευχαριστώ πολύ και για να κλείσουμε τη συζήτηση θα δώσω και πάλι το λόγο στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ και για τη σημερινή σας συμβολή σε αυτή την έκθεση. Όχι, όχι, λειτουργεί, είναι αναμένο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα σημερινά σας σχόλια. Επίση, Επίσης ήταν πολύ αποτελεσματική και ανοιχτή η συνεργασία που είχαμε τους τελευταίους μήνες και έτσι ελπίζω πως στη διάρκεια των επόμενων ημερών θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις τρεις συμβιβαστικέ που ε, παραμένουν κάπως ακόμα ανοιχτές. και που είναι πράγματα τα οποία έχουμε δει και έχουμε συζητήσει και στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ τους όδες τους εκπροσώπους της Κομισιόν και όλους όσοι συνέβαλαν σε, αυτήν την, αυτό το σχέδιο έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And now Mr. Faria for the Committee. Και τώρα ο κύριος Φαρία από την Επιτροπή ΕΜΒ. Εν, μάλιστα, εγώ θέλω μόνο να πω ότι ε, ξενόματος της κυρίας Πιετικάινεν που δεν μπορούσε, που είναι απούσα σήμερα ε, από την αρχή, να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην σύνταξη της έκθεσης και η εργασία μας δεν θα τελειώσει εδώ. Σίγουρα μπορούμε να βασιστούμε στο ΕΛΚΑ για την προώθηση την, ε, του, της υπόθεσης αυτής, του φακέλου αυτού. Και τώρα, Πρόεδρος, να σας θυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο στα διάφορα και μπορούμε να κλείσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση εδώ. Να σας θυμίσω, η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου το απόγευμα και στις 24 το πρωί και το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας όρεξη.